Συνάδελφοι, ο κύριος Έλμερ ζήτησε το λόγο για διαδικαστικό. Κύριε Πρόεδρε, η πρώτη παρέμβαση που έγινε ποτέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από εκλεγμένο Ευρωβουλευτή ήταν από τον ε, Επίσκοπο Dr. Impaisley το 1979 που επέστρεψε το γεγονό ότι η Βρετανική σημαία ε, ήταν κρεβασμένη ανάποδα. Ε, και το 1999 ε, η πρώτη μου παρέμβαση ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο είχε. Σήμερα το πρωί έφτασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γύρω 7 το πρωί και, και πάλι η Βρετανική σημαία κοιμάτιζε ανάποδα. Βέβαια διαπίστωσε ότι στο μεταξύ διορθώθηκε. Αλλά διαβεβαιώστε με παρακαλώ ότι δεν θα επαναλήφθει αυτό το φαινόμενο. Μετά από 33 χρόνια θα έπρεπε να έχουμε μάθει επιτέλους ποια είναι η σωστή φορά για να κρεμάμε την Βρετανική σημαία. It's, um, a failing on the part of the French, I'm afraid. Um έκαναν αυτό το λάθος. Ο κύριος Τσούλορ. Mr. Tudor. Mr. Tudor, you have the floor. Mr. President, may I speak? Yes. Ο κύριος Τσούλορ. Σε ό,τι αφορά το σχόλιο του κυρίου Χέλμερ. Λίγη ησυχία παρακαλώ, λίγη ησυχία. Διαδικαστικό του κυρίου Τιούντορ. Όπως ξέρετε, στην Ευρώπη έχουμε δερμήτα το χειμώνα. Καθημερινά ε, οι πολίτες μας ε, χάνουν τη ζωή τους. Μέχρι στιγμή στη χώρα μου έχουν χάσει τη ζωή τους 75 άνθρωποι. Πραγματική τραγωδία. Σας παρακαλώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε να προτείνετε να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή ε, στη μνήμη των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης από τα δερμήτα το χειμώνα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπάτεν, διαδικαστικό επίσης. Να προσθέσω σε αυτά που είπε ο κύριος Χέλμερ. Ε, είναι ε, γνωστό στον κύριο Χέλμερ ότι ε, όταν η σημαία κυβετίζει ανάποδα δείχνει ε, μια δυσφορία ή μια θλίψη. Νομίζω ότι δεδομένου των καιρών καλύτερα είναι να συνέχεια να αναρτάται με αυτόν τον τρόπο, ανάποδα, λόγω της γενικής ε, θλίψης. Καλώς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόταση. Περνάμε στις ψηφοφορίες τώρα. <clears throat> η ε, γραπτή δήλωση των κυρίων ε, ε, Έντεγκερ Μέγερ για την επιστροφή της του της κατοίκους της έχει υπογραφεί από την πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ζασάντα για να